Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind. Έχετε λάβει τα εγκεκριμένα um, κείμενα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει για τα πρακτικά. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά ούτω. Και τώρα περνάμε στι ε, βάσου του άρθρου